Uh, Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε και σιγά σιγά έρχονται και οι υπόλοιποι, αλλά για αυτού που είναι παρόντες στην ώρα τους, ας αρχίσουμε. Έγκριση μερίσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται. γλώσσε και ανακοινώσει του Πρόεδρου. Δανέζικα, λετονικά και κροατικά δυστυχώς δεν θα έχουμε στη συνεδρίασή μα σήμερα. Τώρα στις 2 Δεκεμβρίου 11 με 12 και 30 στην αίθουσα Γιάννα 6Q2 θα έχουμε μία συνάντηση από κοινού με την Επιτροπή Γυναικών και τη Λίμπε τη δικιά μας όσον αφορά ε, τα θέματα εμπορίας ανθρώπων. Θα είναι συζήτηση αυτή μαζί με την συντονίστρια Μαρία Βασιλιάδου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων και θα μιλήσουμε μαζί της για την έκθεση που αφορά το 2012 με 2016, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την περίοδο δηλαδή. Εκτός μικροφώνου κάποια παρέμβαση. Δεν υπάρχουν γερμανικά, η γερμανική μετάφραση δεν υπάρχει. Αναρωτιέται ο Πρόεδρος. Τώρα είναι εντάξει. Δεν ακούτε γερμανικά. Μα αγγλικά είναι τόσο τέλεια τα αγγλικά σας. Εντάξει τώρα. Okay. It's okay. Είναι εντάξει τώρα, από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Το είχαμε πει και νωρίτερα για τον... τη συνάντηση αυτή με τη συντονίστρια. Σημείο 3 τώρα. Έγκριση πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Και περνάμε στην ημερήσια διαταξή μας αυτή καθε αυτή, στα κυρίως θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του νόμου την ε, συνεργασία και την κατάρτιση στο τομέα αυτό. Έχει να κάνει με τι αποφάσει 2009 2009-371. Η συγκητής μας είναι ο κύριος Δία Δεμέρα και σκιώδης εισηγητές ο κύριος Βάιντενχολτς, ναι, ο κύριος Βάιντενχολτσερ, Κίρκοπ, Πέτερσεν, Έρνστ, Τερικάμπρα και Φεράρα. Θα σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή σε αυτό το θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί ο κύριο Δία Δεμέρα δεν είναι εδώ. Ε, Ακριβώ γι' αυτό σας ε, παρουσιάζω εγώ το θέμα. Και μετά, αν έχετε σχόλια, παρακαλώ. Λοιπόν, βάσει του άρθρου 73 παράγραφος 4 και προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, μετά από κάθε τριμερή διάλογο η διαπραγματευτική ομάδα έρχεται και αναφέρει τι έγινε στην, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Για το θέμα της Europol υπήρξε τριμερής διάλογος στις 18 Νοεμβρίου. Επειδή λοιπόν ο κύριος Διαθεμέρα δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, σας ενημερώνω εγώ βάσει των σημείων που μας παρέδωσε. Τρία θέματα συζητήθηκαν. Πρώτα απ' όλα η συνεργασία μεταξύ χωρών μελών και Europol όσον αφορά την ε, κυβερνητική της δομή για το πρώτο θέμα που καλύπτεται από τα άρθρα 5 έως 8 συζητήθηκε το θέμα επιπλέον διατάξεων για τη συμμετοχή της Europol στην ε, κοινή, σε κοινέ ερευνητικές ομάδες, το ρόλο της Europol και της Eurojust στην, ε, ε, στο ξεκίνημα νέων ποινικών ερευνών και τη δυνατότητα της Europol να έχει απευθείας επαφές με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά τώρα τα θέματα που καλύπτουν τα άρθρα 12 και 22, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη για πρόσθετη αξία του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει εκπροσώπους ως παρατηρητές στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη σύνθεση και την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίση και τι διαδικασίε για τον ορισμό του εκτελεστικού διευθυντή. Όλα αυτά τα θέματα ε, έχουν να κάνουν με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και είναι πολύ σημαντικά για μα. Ο επόμενος τεμερή διάλογος θα λάβει χώρα 8 Δεκεμβρίου και θα ασχοληθεί με θέματα ε, πάλι διατάξεων σχετικά με την διακυβέρνηση και διατάξεων σχετικά με τον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σχόλιο, παρατηρήσεις. Καλώς. Συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο. Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την συνεργασία σε θέματα ποινική δικαιοσύνη. Eurojust. Πάμε πολύ γρήγορα, βλέπω, λέει ο πρόεδρο. Εδώ ο εισηγητή είναι ο Άξελ Φως. Δεν θα κάνω εγώ καμία εισαγωγή. Θα σας δώσω το λόγο ευθύ αμέσω. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Στις 17 Ιουλίου ε, του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση, νομοθετική πρόταση κανονισμού για την Eurojust που περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για την ε, Ευρωπαϊκή για την σύνδεση της Eurojust με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και το ερώτημα προκύπτει είναι γιατί χρειάζεται μεταρρύθμιση η Eurojust. Καταρχάς, ε, Υπάρχει το θέμα της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή ε, Εισαγγελία για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, το οποίο έχει πραγματικά αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια και γι' αυτό προέκυψε και αυτή η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η, εγκλημα, η μορφή εγκληματικότητας, οργανωμένο έγκλημα, συνδέεται με διάφορες μορφές εγκληματικότητας, με διακίνηση ανθρώπων, με εμπόριο ναρκωτικών και... Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ευέλικτη αντιμετώπιση με μονάδες οι οποίες μπορούν να δράσουν διασυνοριακά και ταχύτατα. Χρειαζόμαστε ένα είδους, ε, έναν τρόπο για να αντιμετωπίσουμε διασυνοριακά και πανευρωπαϊκά το οργανωμένο έγκλημα. Η Eurojust δημιουργήθηκε το 2002 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Από την άλλη πρέπει λοιπόν να συνδεθεί. Υπήρξε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο παρουσίασα τον Απρίλιο που μας πέρασε και εδώ σε αυτό το έγγραφο υπήρχαν ορισμένα ερωτήματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εδώ χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση για το τι αρμοδιότητες έχει η κάθε ε, υπηρεσία. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαχωρίσει τις αρμοδιότητες Eurojust και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δίνοντάς τους σαφέστερους ορισμούς. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής εισαγγελία είναι κάτι που φαίνεται πάρα πολύ στο κείμενο και έχει άμεση σχέση με την ε, μεταρρύθμιση της Eurojust. Όπως είπα, τονίζουμε την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και την περασμένη εβδομάδα έγινε συνεδρίαση των σκιωδών συντονιστών κατά την οποία συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της Eurojust, διότι δεν χρειάζονται μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Eurojust. Χρειάζονται μερικές τροποποιήσεις, μερικές ευελτιώσεις, όμως το ζητούμενο είναι η βελτίωση της συνεργασίας, όπως είπαμε, μεταξύ της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χρειάζεται λοιπόν ρύθμιση στον τομέα αυτό Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως ε, δεν έχει νόημα να προχωρήσουμε στην μεταρρύθμιση της Eurojust προτού εξετάσουμε τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό λοιπόν διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την ε, Eurojust μέχρι να δοθούν διευκρινήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι επίσης σημαντικό να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουμε θέσει στο έγγραφο εργασία σχετικά με την μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Γι' αυτό λοιπόν, καλό είναι να κληθεί και το Συμβούλιο να απαντήσει για τη θέση του όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θέλουμε να διοργανώσουμε μία ακρόαση τον Ιανουάριο για όλο αυτό το πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως δεν πρέπει να βιαστούμε, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα οριστεί η συνεργασία των δύο αυτών οργανισμών. Πιστεύω λοιπόν πως η βιασύνη δεν θα μας ωφελήσει το αντίθετο. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό να περιμένουμε. Αυτά ως μια συνοπτική εισαγωγή. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να πω εξ αρχής ότι αρχίσατε τις εργασίες σας την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία. Είπατε να ακούσουμε το Συμβούλιο και το Σκιώδης. Όμως να δώσουμε πρώτα το λόγο στην Επιτροπή. Μετά στο Συμβούλιο και μετά στο Σκιώδης, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και μετά το Συμβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Με τα χαρά να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ήδη ο εισηγητή ανέφερε την ουσία τη ε, πρόταση τη Επιτροπής. Βεβαίω, θέλουμε να βελτιώσουμε την λειτουργία τη Eurojust, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ε, αργαστή συνεργασία μεταξύ τη Eurojust και τη Ευρωπαϊκή Αγγελίας στο μέλλον. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί εκτενώ ε, και στη συνεδριά του Συμβουλίου και θεωρούμε ότι ε, αυτό το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεων. Θα ακούσουμε λοιπόν και από το Συμβούλιο ότι έχει φύγει από την μερική γενική προσέγγιση ε, που θέλει, στην οποία θέλει να καταλήξει το Συμβούλιο σύντομα. Από πλευρά μα έχουν προχωρήσει καλά τα πράγματα, συνεργαστήκαμε με την Ιταλική Προεδρία, ωστόσο θεωρούμε ότι παραμένουν κάποια ζητήματα στο προσχέδιο τη γενική προσέγγιση που μα προβληματίζουν για παράδειγμα, δεν υπάρχει εκπρόσωπο τη Επιτροπή ε, στην τρέχουσα σύνθεση τη Επιτροπή. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. όπως γίνει παλαιότερα στο παρελθόν, το 2012, μετά για το πεδίο εφαρμογή των αρμοδιοτήτων, οριοθέτηση των ε, αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να διευκρινιστεί. Υπάρχει και νέος ε, μηχανισμός ε, αποζημίωσης για τα κατάμελη, όταν υπάρχει διορισμός προέδρου ή αντιπροέδρου. Που, κίνηση με την οποία εμείς διαφωνούμε όμως και έχουμε κάνει και κάποιες προτάσεις να αυξηθεί η επιχειρησιακή λειτουργικότητα της Eurojust με την υποχρέωση ενημέρωσης προς ε, τον οργανισμό. Δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη με την Επιτροπή, επομένως θα επανέλθουμε στο μέλλον. Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ. thank you. And then the presidency, please. Ευχαριστώ, η Πρόεδρε, παρακαλώ. Grazie. Grazie, signor Presidente. Ε, buongiorno a tutti. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και στον εισηγητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που παρουσίασε πολύ ξεκάθαρα την κατάσταση. Η Ιταλική Προεδρία θα φέρει το κείμενο της ε, Eurojust ή μάλλον ένα σημαντικό τμήμα της πρότασης κανονισμού στην ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου ε, Δικαιοσύνης και Αστερικών Υποθέσεων για την μερική γενική προσέγγιση. Συνήθως όταν μιλάμε για τη μερική γενική προσέγγιση αναφέρουμε κάποια περιορισμένα τμήματα του κειμένου. Σε αυτή την περίπτωση όμως το κείμενο είναι σχεδόν πλήρες. και μόνο κάποια τμήματα για την ε, δομή της προστασίας θα μείνουν εκτός του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, γιατί πρέπει να τα εξετάσουμε σε τεχνικό επίπεδο. Όπως και η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτό είναι για τεχνικούς και μόνο λόγους, γιατί η συζήτηση για το θεσμικό επίπεδο, όπως ε, θα εξηγήσει και ο πρόεδρο ε, τη ομάδα εργασία. Οι διαπραγματεύσει λοιπόν συνεχίζονται και γι' αυτό πρέπει κάποια ζητήματα που εκκρεμούν να επιληθούν πριν περάσουμε σε μια συγκεκριμένη δομή συνεργασία μεταξύ τη Eurojust και του Γραφείου τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη δική μα περίπτωση έχουμε ένα πολύτιμο εργαλείο που έχει βελτιώσει το εφιστάμενο σύστημα Eurojust. Είναι πλήρε λειτουργικό και επιχειρησιακό αυτό το οικοδόμημα, μια απόλυτη επιτυχία και κατά τη γνώμη μας με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω η λειτουργία του. Με την εισαγωγή βάσει και του πνεύματος της πρώτης επιτροπής κάποιων τροποποιήσεων σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της Eurojust και ε, την επιχειρησιακή της ικανότητα. Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι θα διατηρήσουμε αυτή τη διτή ε, δομή από πλευράς ε, διοίκησης με την εισαγωγή ενός, ε, μιας εκτελεστικής επιτροπής που θα επιτρέψει ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο να ε, επικεντρωθεί στα επιχειρησιακά. Το βασικό ήταν ένα βασικό αίτημα που είχε γίνει από την αρχή της διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τους δικαστές και εισαγγελείς που εργάζονται στη Eurojust, θα έχουν δυνατότητα να λειτουργούν καλύτερα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Τα διοικητικά ζητήματα θα κατανείμονται ε, μέσω μιας διοικητικής ε, δομής με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι θα συμμετέχει απόλυτα και πλήρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ό,τι φορά τη διαχείριση του Eurojust. Εμείς θα υποβάλουμε το κείμενό μας, όπως είπαμε, στο Συμβούλιο Υπουργών του Δεκεμβρίου. Βεβαίως, ως Συμβούλιο θέλουμε να ξεκινήσουμε και τη διαδικασία των ακροάσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ σύντομα θα συμπληρώσουμε και τα τελευταία κομμάτια του κανονισμού και σίγουρα υπάρχει η προστεθεμένη αξία με την ταχύτατη υιοθέτηση αυτού του μέσου για να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί βάσει των ε, νέων ε, διατάξεων του κανονισμού. Ευχαριστώ. Άξελ, θες να επανέλθεις ε, για να κάνεις κάποιες ε, καταληκτικές ε, παρατηρήσεις. Πριν από αυτό όμως, θα κάνουμε ένα διάλειμμα ενός λεπτού γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα με δύο not picking on you, Axel, <laughs> um, breaking into this important ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν για να επιληθούν τα τεχνικά προβλήματα. If we can adjust some technical issues in two of the booths, if we just have a one minute pause, we'll come straight back to the debate, take two of the shadows, and then you can conclude, Axel. Please don't go away. Uh, we, we... Μη φύγεις, παρακαλώ. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε μεταβίας απαρτία again Διάλειμμα ενός λεπτού λοιπόν. Colleague, colleagues will be restarting in 30 seconds, barely enough time to get coffee, so please make your way back to your seats. Παρακαλώ καθίστε και πάλι στις θέσεις σας για να ξαναξεκινήσουμε. Okay, colleagues, the, um, the issues have been fixed. Ωραία.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 Axel, when you're ready. Axel. Okay. Okay, um... Ωραία. Σίλβι Ιβόν, από πλευρά σοσιαλιστών, από τους Κιώδης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα μεγάλη προσοχή τα όσα υπόθηκαν και καταρχάς θα ήθελα να πω στον εισηγητή ότι συμμερίζω με την άποψή του για το τι έγινε στην συνεδρία των σχεδόν εισηγητών. Πραγματικά πιστεύω πως πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά και να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή όλες τις λεπτομέρειες του φακέλου. Ε, από την άλλη να πω ότι εξακολουθεί να με εκπλήσει το γεγονός ότι μιλάμε για μεταρρύθμιση παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ε, Eurojust. Αυτό προβλεπόταν για τον Δεκέμβριο του 2008. Δεν έχει γίνει όμως και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα όπου συζητούμε για τη μεταρρύθμιση της Eurojust. Και για μένα είναι λίγο δυσνόητη αυτή η διαδικασία μεταρρύθμισης χωρίς πρώτερη αξιολόγηση. Ίσως λοιπόν αυτό θα πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη προσοχή. Το δεύτερο πρόβλημα που θα ήθελα να εντοπίσω εδώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτός ο κατάλογος των αρμοδιοτήτων που προβλέπεται για την Eurojust, ιδιαίτερα το άρθρο 3 παράγραφος 1. Ε, εκεί αναφέρεται η εγκληματικότητα βαριάς μορφής, ενώ στον παλιό κανονισμό αυτός ο κατάλογος αρμοδιοτήτων ήταν ίδιος με εκείνον της Europol. Και εγώ πραγματικά θα ήθελα να μάθω γιατί εδώ αναφέρονται διαφορετικές αρμοδιότητες για τους δύο οργανισμούς. Επίσης, Φυσικά πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ε, σύγκρουσης ε, των αρμοδιοτήτων Eurojust και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να διατηρηθούν οι ισορροπίες. Και τέλος να πω ότι εκπλήσωμαι με το ότι το Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι στο τέλος του χρόνου σκοπεύει να υποβάλει ήδη κείμενο προς εμείς τον Ιανουάριο προετοιμάζουμε μία ακρόαση, όπως υπόθηκε, και πραγματικά ελπίζω η διαδικασία συναπόφασης να τηρηθεί, έτσι ώστε μαζί να συνεργαστούμε για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις της Eurojust. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό η Προεδρία του Συμβουλίου να λάβει υπόψη της την κατάσταση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας. Ευχαριστώ. Ο Λουί Μισελ έχει το λόγο και ο δισηγητής των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η κυρία Γκρισμπέκ δεν μπορούσε να περιβρεθεί σήμερα. Μου ζήτησε λοιπόν να την αντικαταστήσω. Θα σας μεταφέρω λοιπόν τις ε, παρατηρήσεις της. Όσο ασκιώδη εισηγήτρια της Άλντε για το φάκελο της Eurojust, θα στηρίζω την προσέγγιση του εισηγητή μα, κυρίου Άξελ Βος, με τον οποίο συμφωνήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση ε, των σκιωδών, να αναστείλουμε τις εργασίες μας επί του φακέλου ε, μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Συγκυλία. μας φαίνεται μη λογικό και μια κακή χρονική στιγμή να μιλήσουμε τώρα για τη μεταρρύθμιση της Eurojust ε, εν ώψη ε, της νέας, ε, των διαπραγματεύσεων για τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις διαπραγματεύσει για την Eurojust. Πρέπει να περιμένουμε όμως μέχρι το τέλος τους για να περάσουμε σε μεταρρύθμιση μέχρι τη, μάλλον, την οθέτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Πρώτον, πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι δύο φορεί, Eurojust και Ευρωπαϊκή Συγγελία. Ποια θα είναι η έδρα του, θα είναι η ίδια, θα έχουν την ίδια δομή ή θα υπάρχει διτή δομή. Θα ασχολούνται με τα ίδια ζητήματα διαφορετικά. Είναι βασικά ερωτήματα, αλλά υπάρχουν πολλά σημεία προβληματισμού τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε, ούτω ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά οι δύο οργανισμοί μα. Φαίνεται ότι η Eurojust είναι ένα οργανισμό που λειτουργεί αρκετά καλά, από αυτό που μα λένε τουλάχιστον, Όμω, στη Γαλλία, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι από ε, την διαδικασία μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο το 2013 ε, στα 36 εφετία της Γαλλίας, μόνο ένα μετέφερε ε, ενημέρωση προς τη Eurojust. Ποια είναι λοιπόν η λειτουργία της Eurojust. Ξέρουμε ότι λειτουργεί σε θελοντική βάση, αλλά πρέπει αυτό να ενισχυθεί αν θέλουμε να ενισχύσουμε την δικαστική συνεργασία. Με τη Eurojust, την δικαστική συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών και την διαμόρφωση κοινού χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά, για την προστασία δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το διακύβευμα για τη λειτουργία της Eurojust και θα πρέπει να ε, δοθούν τα απαραίτητα εχέγγυα για τα δεδομένα ε, όλων των ε, μερών. Αυτά ήθελα να αναφέρει η Σκιώδης. Ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Άξελ για τα σχόλιά του. Θέλετε? Άξελ, έχετε ερωτήσεις? Υπάρχει χρόνος. Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις προς το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, μπορείτε και αργότερα, αλλά και τώρα, αν θέλετε, παρακαλώ τις τελικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντ. Καταρχάς, όσον αφορά την ε, διπλή δομή, φυσικά και πρέπει να δούμε αυτό το θέμα πάρα πολύ προσεκτικά και να μην λάβουμε βιαστικές αποφάσεις, διότι πρόκειται για έναν οργανισμό πάρα πολύ σημαντικό και ίσως είναι συνετό αυτή η εθελοντική βάση εργασίων του Eurojust να συνεχίσει. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση της Eurojust. Ε, εδώ να πω ότι η συνάδελφος κυρία Κάουφμαν έχει απόλυτο δίκαιο. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από ό,τι ακούω όμως, η αξιολόγηση έχει ήδη ολοκληρωθεί και το πόρισμα δεν ήταν και ιδιαίτερα διαφορετικό από τα συμπεράσματα που είχαμε βγάλει έτσι και αλλιώς. Θα ήθελα επομένως να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους και οδησηγητές για τον ρεαλισμό που έδειξαν. Γιατί πραγματικά χρειάζεται να δούμε πώς η συνεργασία ανάμεσα στην Eurojust και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βελτιωθεί. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε και να διορθώσουμε σε τελικό στάδιο. Φυσικά είναι κάτι που θα διαρκέσει κάποιο χρόνο, ιδιαίτερα όσο περιμένουμε το Συμβούλιο να ολοκληρώσει τις εργασίες του και μετά να περάσουμε στη διαδικασία των τριμερών διαλόγων. Άξελ, είναι σαφές. Έχετε καταδείξει και εσύ και οι σκιώδεις εισηγητές τα ζητήματα του τριμερή Διαλόγου. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να δώσουμε το λόγο ξανά στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Έχουν εντοπιστεί τα ζητήματα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Νομίζω ότι απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εμείς. Αν δεν θέλει κανείς άλλος το λόγο για ερωτήσεις στην Επίτροπη το Συμβούλιο, συνεχίζουμε. Η κυρία Μακοβέη δεν είναι εδώ που είναι υπεύθυνη για το επόμενο θέμα, οπότε είναι πρακτικό το ζήτημα τι κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, δεν νομίζω. Το τελειώσαμε. Η κυρία Μακοβέη δεν έχει έρθει. Ξέρουμε τι ώρα θα έρθει. Προσπαθούμε να την εντοπίσουμε. Συγγνώμη συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε με το επόμενο θέμα. Αυτό θα πει να είναι κανεί καλός πρόεδρος. Προχωράει πολύ γρήγορα με την ημερήσια διάταξη. Αλλά το τίμημα τη επιτυχία αυτή είναι ότι να δεν έχουμε τον επόμενο συνάδελφο εδώ. Τηλεφωνάμε στο γραφείο της για να δούμε. Αλλά θα διακόψουμε στο μεταξύ για λίγο. Πολύ γρήγορα θα σας πω. Όποτε καταλαβαίνω έρχεται.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 Colleagues, uh, Mrs. McAvey has entered the room. Μόλις μπήκε στην αίθουσα κυρία Μακοβέη, αγαπητοί συνάδελφοι. Okay, uh, Συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Ήρθε η κυρία Μακοβέη, οπότε περνάμε στο θέμα της υπηρεσίας του Ευρωπαίου Εισαγγελία. Ξέρετε ότι τον Ιούλιο είχαμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δημιουργηθεί η υπηρεσία αυτή βάσει του άρθρου 86 της Συνθήκης συμφωνήθηκε από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, ήρθε η πρόταση για σύμφωνη γνώμη στο Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται για συναπόφαση, πρόκειται για σύμφωνη γνώμη, έτσι. Πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτό συνάδελφοι. Εμείς εγκρίναμε ψήφισμα, θα το θυμόσαστε ίσως ότι ήταν εισηγητής ο κύριος Ιακολίνος στην προηγούμενη θητεία μας βάσει του άρθρου 81 του κανονισμού με πράγματα που λέγαμε στο Συμβούλιο για τη μορφή που πρέπει να έχει η υπηρεσία αυτή και πώς θα έπρεπε να εργάζεται. Και ζητήσαμε από το Συμβούλιο να εμπλέξει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερα το να συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα έχουμε λοιπόν την Επιτροπή του Συμβούλιο για να μας ενημερώσουν ε, το νέο εισηγητή για την υπόθεση αυτή, την κυρία Μακοβέ, οπότε θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά στην Ιταλική Προεδρία και μετά στην εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές, για να ακούσουμε τη γνώμη τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα, που εκπροσωπείται από τον κύριο Χάβετ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευθύ αμέσω, παρακαλώ, για να μας ενημερώσει σύντομα για την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αρχίζω λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τι προσπάθειε τη Ιταλική Προεδρία να προχωρήσει παρετέρω όσον αφορά τι διατάξει και συμμετέχουμε επικοδομητικά στη συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι το επίπεδο προστασίας και συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το ίδιο όταν πρόκειται για πάτε σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία του κοινοτικού προπολογισμού είναι κοινό ο στόχος και η υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο, την προστασία δηλαδή των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το να υπάρχει ένας ανεξάρτητος Ευρωπαίος Αγγελέας το 2016 είναι μια επιθυμία η οποία επιβεβαιώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία αποτελεσματική και αποδοτική ευρωπαϊκή συγγελία. Και αυτέ είναι οι κόκκινε γραμμέ μα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι ανεξάρτητη υπηρεσία αυτή. Μακριά από πολιτικέ επιρροέ, αλλά να λογοδοτεί για το έργο τη ο εισαγγελέα, οι αναπληρωτές και όλοι οι αξιωματούχοι πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους. Βέβαια, η διαδικασία ορισμού πρέπει να προβλέπει ακριβώς τη δυνατότητα και την, ε, να διασφαλίζει ουσιαστικά την ανεξαρτησία των ατόμων αυτών. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε την επιλογή μεταξύ διαφορετικών ε, υποψηφίων. Χρειάζεται εμπειρία, γνώση που να αξιολογείται από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε τοπικό επίπεδο οι εξουσιοδοτημένοι εισαγγελίε που δρούν εκ μέρου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα βρίσκονται μακριά από το κέντρο, αλλά πρέπει να έχουν του ίδιου στόχου και να του εφαρμόζουν όσο γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι ζωτική σημασία η ευθύνη να αξιολογείται από ε, μια ενιαία κριτική επιτροπή. Έπειτα, πρέπει η υπηρεσία αυτή να είναι αποτελεσματική. Η κατανομή εργασία στην υπηρεσία πρέπει να επιτρέπει και αυτού που βρίσκονται επί τόπου, του εξοδοτημένου αγγελεί δηλαδή, και εκείνου που βρίσκονται στο, σε κεντρικά γραφεία, να εφαρμόζουν την ίδια πολιτική για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση. Στο σχέδιο ε, αναφέρεται την επιθυμία να υπάρχει μια καλή ισορροπία. Το κέντρο πρέπει να έχει εποπτικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις ε, διάφορες διαδικασίες επιτόπου. Επίσης είναι ζωτική σημασία να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων, χωρίς όμως να παραβιάζονται οι ρήτρε ε, ασφαλείας για τους υπόπτους ή τους κατηγορούμενους. Τα δικαιώματα αυτών πρέπει να γίνονται σεβαστά βάσει και της εθνικής νομοθεσίας. Επίσης, ο κανονισμός αυτός προβλέπει και νέα δικαιώματα για τους υπόπτους, όπως εκείνο των ε, συλλογής αποδεικτικών ε, στοιχείων, με υψηλού επίπεδου ρήτρες διασφάλισης. Επίσης, προτείνει Επιτροπή και μέτρα αναθεώρησης που θα συνοδεύονται από τη δυνατότητα για προδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τέλος, η Επιτροπή θέλει να συνεργαστεί με την νέα συγκεκριτή, την κυρία Μακοβά για αυτό το σημαντικό θέμα. Έχουμε τον ίδιο στόχο, είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών, έχουν ένα σύστημα το οποίο στην πράξη να εφαρμόζεται ικανοποιητικά και να αποτελεί μια πρόσθετη αξία στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλαζάρ, τώρα εκ μέρους της Προεδρίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μακοβέη. Πριν από οτιδήποτε άλλο θα ήθελα παρακαλώ να επιμείνω στο εξή. Εμείς ανταποκρινόμαστε στην πρόσκληση που μας έγινε στα πλαίσια της έκθεσης Ιακωβίνο στην προηγούμενη θητεία. Δηλαδή ότι θέλουμε και εμείς πράγματι να ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο. Είπατε και εσείς ότι πρόκειται για μια ειδική διαδικασία γιατί δεν είμαστε σε συναπόφαση αλλά ο Ιταλός Υπουργός θέλει να εμπλέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται περισσότερο στην υπηρεσία αυτή της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Στην Ιταλική Προεδρία η συζήτηση για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα αποτέλεσε αντικείμενο δύο συζητήσεων ε, σε υπουργικό επίπεδο. Θα είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Τζάι του Δεκεμβρίου στην άτυπη συνάντηση που θα έχουμε στο Μιλάνο. Ο κύριος Λάντον ε, στο θέμα των διαδικαστικών εγγύσεων. Δηλαδή στον ε, έλεγχο των ε, πράξεων του Ευρωπαίου Εισαγγελέα βάσει της δικαιοδοσίας. Όλα αυτά συζητήθηκαν στο Συμβούλιο τον Οκτώβριο και αυτό που βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεων είναι ο χώρος ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Ποια είναι η δικαιοδοσία δηλαδή βάσει της οποίας ο Ευρωπαίος εισαγγελέα θα μπορεί να εργάζεται ως ενιαίος ε, εισαγγελέα που θα ερευνά τις, ε, τα επιμέρους αδικήματα. Είναι επίσης κάτι το οποίο συζητήσαμε και στις τέσσερις συνεδριάσεις που είχε η Επιτροπή η οποία ασχολείται με τα ποινικά ζητήματα, το CTS. Προχωρήσαμε λοιπόν στα βασικά στοιχεία της συζήτησης αυτής. Ιδιαίτερα συζητήσαμε το ζήτημα της δομής, εννοείται. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η προηγούμενη Προεδρία μας άφησε ένα κείμενο αρκετά προχωρημένο και αρκετά διαρθρωμένο όσον αφορά την δομή του σώματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι πράγματα τα οποία βρήκαμε από την προηγούμενη Προεδρία. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τα κύρια ζητήματα και τα πιο σημαντικά που παραμένουν σε κρεμότητα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες διαπραγματεύσεις εκ παραλλήλου. Συζητήσαμε λοιπόν, προχωρήσαμε στο θέμα των ερευνών που κάνει ο εισαγγελέα. Ποια είναι η μέθοδος των ερευνών που γίνονται από περισσότερες από μία χώρες. Ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στις εξουσίες του εξοδοτημένου εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των εξουδετημένων αυτών εισαγγελέων. Έπειτα πώς θα γίνεται ο δικαστικός έλεγχος από τις εθνικές αρχές όταν πρόκειται για την εφαρμογή ερευνών και διεξαγωγή μάλλον ερευνών από μία χώρα στη άλλη. Έπειτα, πώς γίνεται η καταχώρηση των διαφόρων περιπτώσεων που υποβάλλονται στον εισαγγελέα. Βάσει του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ότι αυξάνουμε σημαντικά τον ε, έλεγχο όσον αφορά τη δικαιοδοσία των ε, πράξεων που είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Συζητήσαμε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία και συζητήσαμε και τις εγγύησεις για τους υπόπτους κατηγορούμενους. Στο άτυπο, στην άτυπη συνάντηση του Μιλάνου, οι Υπουργοί, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπάθησαν να ενισχύσουν όσο γίνεται περισσότερο τα δικαιώματα των ατόμων τα οποία μπλέκονται σε διαδικασίες οι οποίες, τις οποίες αναλαμβάνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Και είπαμε ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να ισχύουν σε όλες τις χώρες που εμπίπτουν σε αυτή τη δικαιοδοσία. Αναφερθήκαμε επίσης στα δικαστήρια τα εθνικά. Είπαμε ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από τις εθνικές αρχές και είπαμε επίσης ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Δεν το έχουμε αποφασίσει όμως ακόμα. Συνεχίζουμε να το συζητάμε και εξετάζουμε τη δυνατότητα απευθείας ε, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε κάποιες ειδικέ περιπτώσεις. Επιμένω όμως ότι η συζήτηση συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει και το θέμα της προστασίας δεδομένων. Αυτό όμως συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζουν, συνεχίζονται. Αναφερθήκαμε και στο προσωπικό. Το ερώτημα που τέθηκε είναι ποιο θα είναι το καταστατικό των μελών της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Με ποιο καθεστώς θα δουλεύουν. Υπάρχουν Ευρωπαίες Αγγελίες, οι οποίοι προέρχονται από όλες τις χώρες μέλη. Θα ανήκουν στην εθνική δικαιοδοσία ή θα έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς, θα είναι προσωρινή υπάλληλοι, ας πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, κάποια ζητήματα που εξετάσαμε. Συζητήσαμε και για τις σχέσεις με τους εταίρους, με τη Eurojust. Η σύνδεση με τη Eurojust είναι κάτι ζωτική σημασίας. Όσον αφορά τις έρευνες που έχουν να κάνουν με κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Εάν υπάρξει τέτοια ενισχυμένη συνεργασία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έτσι καλώς δεν συμμετέχουν γιατί αποκλείονται από τον τίτλο 5 της συνθήκης. Η διαβίβαση δεδομένων τώρα. Το Δεκέμβριο είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε κάποια άρθρα τα οποία ελπίζω να πετύχουν ευρεία συνένεση. Ήδη συζητάμε για την προσφυγή στη δικαιοσύνη, άρθρο το οποίο θα είναι υπό την ευθύνη της Προεδρίας και μόνο. Επίσης, θέτουμε στον Υπουργό και ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το καθεστώς και την ανεξαρτησία των εθνικών ε, μελών αλλά και του Γενικού Εισαγγελέα. Μπορούμε να φανταστούμε ένα σύστημα το οποίο συζητιέται και συζητιόταν και στην προηγούμενη θητεία και που έχει να κάνει με την ανεξαρτησία του Γενικού Εισαγγελέα και επ' αυτού θα γίνει πρόταση. Έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες αποστάσεις από τον ορισμό από τις χώρες μέλη και να προτιμήσουμε αυτούς που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, οι οποίοι θα μπορούν έτσι να είναι υποψήφοι. Φυσικά θα υπάρξει μια ομάδα που θα κάνει την επιλογή, που θα επιλέξει τους μεταξύ των υποψηφίων αυτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα μπορεί να αποφανθεί από αυτού. Αυτή είναι η κατάσταση συζητήσεων σήμερα στο Συμβούλιο. Θέλουμε πράγματι να καταλήξουμε σε μία απόφαση η οποία να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της ε, Γενικής Αυτής Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ με τα βήματα που κάνει η Προεδρία. Τώρα για να ολοκληρώσουμε θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιταλική Προεδρία για το ότι ασχολήθηκε με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σχετίζεται με το ψήφισμα του Μαρτίου, στο οποίο το Κοινοβούλιο ζήτησε να εμπλακεί ενεργά στις ε, διαβουλεύσεις. Το θέμα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, η διαδικασία επίσης, και γνωρίζουμε ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα στο Συμβούλιο. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε μια ξεκάθαρη θέση όσον αφορά την δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ελπίζουμε να γίνουν και κάποιες υποχωρήσεις από το Συμβούλιο σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα μπορέσει να απαγγέλει κατηγορίες και να οδηγεί στο δικαστήριο όσους παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ευρωπαϊκής Δικαστικής Συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κάτι διαφορετικό από την Eurojust και έτσι πρέπει να παραμείνει. Και οποιαδήποτε λύση που δεν θα οδηγήσει σε βελτίωση της Ευρωπαϊκής ευαγγελίας δεν πρέπει να γίνει δεκτή ούτε για τους φορολογούμενους ούτε και για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Σε αυτό το στάδιο το Συμβούλιο βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία σχεδιασμού και πρέπει να δοθεί προσοχή, όπως τόνισα, στην ανεξαρτησία. Γνωρίζουμε την επιθυμία του Συμβουλίου για την ε, δομή, τη διοικητική δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εμείς πιστεύουμε ότι η δομή αυτή είναι σωστή, ωστόσο οι εξουσίες πρέπει να διατηρηθούν σε κεντρικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ανοιχτή διαδικασία διορισμού των εισαγγελέων και αυτό θα γίνει μόνο με προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού και αξιολόγηση των υποψηφίων από μια κριτική επιτροπή εμπειρογνώμων με συμμετοχή φυσικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε μία δομή με μέλη όπως της Eurojust, τα οποία διορίζονται, αλλά μέλη τα οποία θα προσλαμβάνονται με διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού. Η δομή του εισαγγελικού σώματος θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και εμείς προτείνουμε μία εξειδίκευση των διάφορων σωμάτων της εισαγγελία ανάλογα με τα αδικήματα και όχι ανάλογα με την εθνικότητα. Διότι διαφορετικά θα διακυβευτεί η ανεξαρτησία όσον αφορά τις ε, υποθέσεις που θα εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης, χρειάζεται μία πιο ε, σαφής αναφορά των αρμοδιοτήτων. Χρειάζεται όχι μόνο έλεγχος και παρακολούθηση των υποθέσεων, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να αναλάβει και ηγετικό ρόλο στις διασυνοριακές ε, εκδικάσεις ποινικών ζητημάτων. Ταυτόχρονα, η διπλή λύση για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς μπορεί να είναι μόνο αποτελεσματική εφόσον δεν επηρεάζεται η ανεξαρτησία των ε, εισαγγελέων. Όσον αφορά τώρα το παραδεκτό των αποδείξεων, εμείς προτείνουμε κάποιες ε, καινοτόμες λύσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί, βελτιωθούν οι συνθήκες στην ε, ποινική δικαιοσύνη. Προτείνουμε μία εναρμόνιση της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους ε, σκόπελους της ε, διασυνοριακής συνεργασίας. Ιδιαίτερα στο θέμα της ενομικής αρρωγής, τις διασυνοριακές υποθέσεις, χρειάζεται εναρμόνιση των, της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και της δικαστικής συνεργασίας ανάμεσα στις αγγελικές αρχές κρατών μελών. Γι' αυτό χρειάζονται τα κατάλληλα νομικά μέσα τα οποία θα διευκολύνουν τη συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις. Χρειάζεται επίσης να διωθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ασφαλιστικές δικλίδες που θα προστατεύουν τους υπόπτους και τους κατηγορουμένους. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα. Όσον αφορά τώρα την δικαστική, το δικαστικό έλεγχο, χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα προσφυγής. Και χρειάζεται να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αποτραπεί η τεχνητή παρεμπόδιση της δικαστικής διαδικασίας. Συμπερασματικά λοιπόν χρειάζεται μία δομή που να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και ελπίζω οι επερχόμενες προεδρίες να συνεχίσουν την καλή συνεργασία μαζί μας. Και καλό το Συμβούλιο να συμπεριλαμβάνει πάντοτε το Κοινοβούλιο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και να δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να δώσει την τελική του έγκριση στη σύσταση αυτού του νέου οργανισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η ε, Μπριγκίτα έχει το λόγο. My apologies. Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία για μένα παραμένουν άλυτα. Και η Προεδρία του Συμβουλίου μας ενημέρωσε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή. Ωστόσο να πω ότι θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των ε, διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο, διότι το τελευταίο κείμενο που μας ε, δόθηκε από το Συμβούλιο μας δόθηκε το Μάιο. Και το κείμενο αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στην δομή της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα παραμένουν και πιστεύω ότι χρειάζεται να ενημερωθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τα επιμέρους ε, άλυτα ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω να μας στείλετε γραπτά τις νεότερες εξελίξεις στο Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να διατυπώσουμε μια εμπεριστατωμένη και συνοπτική και ολοκληρωμένη άποψη. Τώρα θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημαντικά για μένα θέματα. Καταρχάς, όπως είπε και η συγγήτρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τη δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από ό,τι βλέπω από το κείμενο του Μαΐου, βλέπω ότι θα υπάρχει ένα σώμα εισαγγελέων που θα αποτελείται από πολλές από πολλέ δομές και πραγματικά μου φαίνεται κάπως περίπλοκη η δομή του λοιπόν και αναρωτιέμαι εάν θα έπρεπε η δομή να είναι πιο απλή έτσι ώστε να είναι και πιο αποτελεσματική. Για παράδειγμα, στην πρόταση αυτή αναφέρεται ένα σύστημα όπου κάθε τρία χρόνια θα αλλάζει το 1 τρίτο των εισαγγελέων. Αλλά πραγματικά ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό θα λειτουργήσει. Δεν καταλαβαίνω το όφελος που θα αποκομίσουμε. Έπειτα, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάτι που αναφέρθηκε έτσι καλλιώς στην αρχή, η ανάγκη δηλαδή για μια πραγματικά ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου μας μίλησε για την ανεξαρτησία του επικεφαλής των ερευνών και είδα τις γνωμοδοτήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και η γνωμοδότηση του Γερμανικού Κοινοβουλίου έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση όσον αφορά της, την ανεξαρτησία, δηλαδή το ότι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής εισαγγελία θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι θα διασφαλίζεται η απόλυτη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Όμως, στο έγγραφο που έχω μπροστά μου διαβάζω κάτι τελείως διαφορετικό. Μία διαδικασία διαφορετική όπου τον ηγετικό ρόλο θα έχει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα έχει απλά συμβουλευτικό ρόλο. Αυτή η πρόταση που έκανε το Γερμανικό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα από εμάς, διότι πιστεύουμε ότι έτσι θα διασφαλιστεί ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έπειτα, ο ορισμός των εισαγγελέων, εδώ αναφέρομαι στα άρθρα 14 και 15 του κειμένου που έχω από τον Μάιο, είναι κάτι που μου δημιουργεί ερωτηματικά. Πραγματικά εδώ δεν προβλέπεται κάποια ανάμιξη των εθνικών εισαγγελιών. Και αυτό είναι κάτι τελείως ε, διαφορετικό από αυτό που έχουμε φανταστεί μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι πώς ακριβώς θα γίνει ο ορισμός των εισαγγελέων από κάθε κράτος μέλος. Τρίτο ζήτημα. Μιλήσαμε για την σύνδεση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Eurojust και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία σύγκρουση αρμοδιοτήτων εδώ ενδεχομένως. Ε, και πέραν αυτών έχουμε και τον Όλαφ ο οποίος συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μάθω από το Συμβούλιο πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Όλαφ, Eurojust και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πιστεύω πως εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο. Έπειτα, στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε αρκετό καιρό πριν, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα πρέπει να επιφέρει και επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω και το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και εκτιμήσεις σχετικά με το επιπλέον κόστος. Και τελευταία ερώτηση. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε ήδη σε αυτό στην αρχή της δίκαιης δίκης. Γνωρίζουμε ότι τα δικονομικά δικαιώματα είναι ακόμα ένα άλυτο θέμα, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μάθω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα των κατηγορουμένων διότι χρειάζεται να διατυπωθούν σαφέστερα. Και αυτό είναι ένα σημείο για το οποίο θα ήθελα να μάθω πολύ περισσότερες πληροφορίες. Και επίσης είδα ότι στο κείμενο του Συμβουλίου, στο άρθρο 5, γίνεται λόγος για διασφάλιση ότι για διασφάλιση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η διατύπωση μου φαίνεται αρκετά αδύναμη. Για ποια θεμελιώδη δικαιώματα μιλάμε. Διότι εδώ πρέπει να αναφέρονται σαφέστατα τα δικαιώματα τα οποία αναφέρει η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και φυσικά η διασφάλιση τους. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άποψη του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ Σίλβια. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξανά για να απαντήσει στις συγκεκριμένες ερωτήσεις της εισηγητρίας. Πριν από αυτό όμως ο Τίμωθη Κέρκοπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ακολουθώ κι εγώ τις παρατηρήσεις της κυρίας Κάφμαν. Όπως ξέρετε και εγώ βεβαίως μιλώ εξ ονόματος ε, των ε, συντηρητικών μεταρρυθμιστών του ECR. Από πλευρά Ηνωμένου Βασιλείου όμως ε, έχουμε κάποιες εμφωλίες για το πρωτόκολλο 21 και, και η Δανία εξαιρείται ε, αυτομάτως ε, από το πρωτόκολλο αυτό και το 22. Το αναφέρω αυτό παρεμπιπτόντως, επειδή από τη σκοπιά της δικής μας ομάδας εμείς ε, στηρίζουμε θερμά οτιδήποτε είναι αποτελεσματικό και λογικό για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της απάτης και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε και καταπολεμήσουμε αυτά τα εγκλήματα. Κυρίως όμως ε, εν είδη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με την αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων και εργαλείων που θεωρούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν αξιοποιούνται παρκώς. Η κυρία Κάφμαν μόλις επεσήμανε κάποιες ε, ε, επιφυλάξεις από πλευρά Γερμανίας και άλλα κράτη-μέλη έχουν Επιφυλάξει για κάποιες προτάσεις. Θα ήθελα να επισημάνω μερικούς από τους τομείς όπου πιστεύω ότι χωλαίνει με κάποιο τρόπο αυτή η πρόταση. Πρώτον, η πρόταση δημιουργεί διαφορετικά συστήματα. Και έτσι δημιουργείται σύγχυση σε ό,τι αφορά την πόλωση ε, για την καταπολέμηση ε, του οργανωμένου εγκλήματος, κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για την καταπολέμηση της ε, φορολογικής απάτης, γιατί ενέχει και συνεπάγεται την προκαταβολή ή και την υποκατάσταση πολλών αρκετά αποτελεσματικών εθνικών πολιτικών. Επομένω, οι διαχωριστικέ γραμμέ μεταξύ αυτής της ε, αποκλειστικής εξουσίας και του υφιστάμενου καθεστώτος θα δημιουργήσει σύγχυση και έτσι θα χάσουμε πολλές ε, πρωτοβουλίες που θα αναλαμβάναμε διαφορετικά. Δεύτερον, νομίζω ότι η εισηγήτρια κυρία Μάκοβέη ανέφερε υψηλό κόστος. Εγώ διαφωνώ. Το αντίθετο μάλιστα αναφέρω. Η Επιτροπή έχει ήδη αναφέρει ένα ενδεικτικό αρχικό κόστος μόλις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και ετήσια, ετήσιο κόστος λειτουργίας ε, που αρχικά είχε εκτιμηθεί στα 20 εκατομμύρια ευρώ και τώρα, χάρη σε περικοπές και εξοικονόμηση που γίνεται από ε, τον προπολογισμό της Eurojust, περνάμε στα 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Με κάθε σεβασμό επειδή έχω κοιτάξει και το κόστος των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τα όσα κάνουμε, αυτά τα, τα ποσά είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που προτείνονται. Αν έχουμε σημαντικές φιλοδοξίες ε, για τους προπολογισμού μας, θα πρέπει να έχουμε ε, μεριμνήσει, ώστε να, τα, να μπορούμε όλα αυτά να τα πληρώσουμε. Είναι πολύ μικρό το ποσό λοιπόν και έτσι μου δημιουργείται η εικόνα ότι η αποτελεσματικότητα ε, τελικά θα είναι πολύ περιορισμένη, ιδίως με τις αποκλειστικές εξουσίες που θα αναλάβει. Να προσθέσω κάτι εδώ. Ισχυρίζονται ότι όχι μόνο το κόστος θα είναι πολύ χαμηλό, αλλά και όλο το υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα της αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων. Νομίζω ότι η κυρία Κάφμαν το ανέφερε προηγουμένως, πώ ακριβώς ε, θα διορίζονται αξιωματούχοι για να εποπτεύουν αυτή τη λειτουργία αυτού του οργανισμού. Είναι ένα ζήτημα εδώ που πρέπει να αποφύγουμε την εθνική ε, κυριαρχία και να έχουμε ε, ανοιχτούς διαγωνισμούς. Όμως αυτό είναι που θα δημιουργήσει σύγχυση και αναποτελεσματικότητα. Αν προσπαθούμε να είμαστε έτσι αντικειμενικοί, έχουμε δει και άλλα θεσμικά όργανα που είναι αποτελεσματικά, γιατί αποφασίσαμε ακριβώς να ψάξουμε και να βρούμε τους ε, πλέον αποδοτικούς ε, υποψηφίους που να έχουν ε, την πλέον κατάλληλη εμπειρία. Και αυτούς διορίσαμε. Βέβαια μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, Βρετανός είστε, αυτό θα πείτε. Αλλά Έχουμε και το παράδειγμα του Ρόμπιν Wright, ε, επικεφαλής της Europol. Ναι, ήταν Βρετανός ε, αστυνομικό, αλλά είχε τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειαζόμασταν για να ηγηθεί ενό ε, τέτοιου αστυνομικού οργανισμού και τον στηρίζουμε πλήρω. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Αν ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική που προτείνεται, νομίζω ότι έχουμε χαμηλότερε πιθανότητε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την αποτελεσματική συνεργασία. Ναι, εντάξει, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, αλλά ανησυχώ ότι και άλλες χώρες, και η Γερμανία, αλλά και άλλες έχουν πολύ αποτελεσματικά συστήματα και ήδη καταπολεμούν αυτές οι κατηγορίες εγκλήματος, ήδη τα διώκουν όπου δει. Και έτσι θεωρώ ότι το να έχουμε ακόμα ένα επίπεδο με τέτοιο είδος αποκλειστικότητας είναι σφάλμα. Τέλος, ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε σίγουρα είναι να συγκεράσουμε τις ε, καλύτερες πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές από όλα τα κρατημέλη, αλλά και να συνεργαστούμε περαιτέρω για το ζήτημα της συνεργασίας, της, ε, του εντοπισμού και της δίωξης. Νομίζω ότι το έχουμε εξετάσει επιφανειακά και μόνο. Έχουμε πολλές τέτοιες εμπειρίες από τις κοινέ ε, ομάδες ερεύνης. Θα θυμάστε, πρόεδρε, ότι και εγώ ήμουν επικεφαλής αυτής της ομάδας για την έκθεση. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ... θεωρούσαμε ότι θα ήταν πολύ θετικά. Τελικά όμως ήταν απογοητευτικά εξαιτία της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ ε, των οργανισμών επιβολής του νόμου. Πρέπει να εργαστούμε με αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Πολλά υπάρχουν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές, ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση, αλλά γιατί να μην το κάνουμε αυτό με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά τους και να τα αξιοποιήσουμε επαρκώς. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μισελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά με τα χαράς ακούω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμμερίζονται αυτή τη βούληση εγκαθίδρυσης ε, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας το ταχύτερο δυνατό. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τίμημα. Γι' αυτό και συμμερίζομαι απολύτως ε, τους προβληματισμούς που ανέφεραν ε, που ανέφερε συνάδελφος Κάουφμαν η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι γνωστή, να την υπερθυμίσουμε. Είχε ψηφιστεί επί της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Και πρέπει να μην ε, απομακρυνθούμε από αυτήν. Πολλοί λένε ότι η Ευρωπαϊκή Συγγελία αποτελεί σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το γνωρίζουμε όλο αυτό. Βεβαίω αυτό άπτεται και τη εθνική κυριαρχία ε, των κρατών μελών και της, ε, των δικαστικών αρχών. Γι' αυτό και θα υπάρχει και η κίτρινη κάρτα ε, για τις εθνικές αρχές. Απαιτείται και απόλυτη νομιμότητα και πλήρη στήριση των ευρωπαϊκών μας αρχών. Αυτή η νομιμότητα λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίζει την στενή συνεργασία μεταξύ των επιμέρους αρχών. Γι' αυτό θέλουμε το Συμβούλιο να εμπλέξει πλήρως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις με τη διοργάνωση κοινών συνεδριάσεων για να υπάρχει εξισορροπημένη εκπροσώπηση των θεσμικών οργάνων. Είναι μια πολύ πιο κατάλληλη και ισορροπημένη προσέγγιση. Βλέπουμε την ε, νέα ε, τροπή που παίρνει η πρόταση της Επιτροπής για τη δομή της εισαγγελία. Νομίζω ότι ε, πλήττει και αποδυναμώνει την νέα σύνθεση. Γι' αυτό, από τη δική μας ομάδα τουλάχιστον, είμαστε υπέρ της ομοσπονδιακής διάρθρωσης και όχι διακυβερνητικής. κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της Ευρώπης. Ε, γιατί θα πρέπει να μεριμνούμε για τα δικαιώματα των πολιτών μας. Και τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να αποδείξουμε ότι θα είναι σε θέση να ε, εγκαθιδρύσουν ε, συστήματα που θα είναι αποτελεσματικά και δίκαια και να μην τροφοδοτούμε εμείς τον ευρωσκεπτικισμό. Δεν θέλω να επανέλθω, αλλά υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που είναι απόλυτα θεμελιώδη. Ε, ο συνάδελφος προηγουμένως αναφέρθηκε στο κόστος. Πρέπει να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό αυτό το κόστος που προτείνει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή. Μπορεί να ακούγεται πολύ ευχάριστο και ελκυστικό. Πρέπει όμως να είμαστε και ρεαλιστές. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει το κόστος να ε, αποτελέσει εμπόδιο σε ένα τόσο σημαντικό βήμα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ευχαριστούμε, Λουί. Γιάν Άλμπερτ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω ότι χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία για να καταπολεμήσουμε τη ζημιά που γίνεται από τα εγκλήματα αυτά σε βάρος της Ευρώπης. Όλοι συμφωνούμε ότι επήγει, γιατί τα νούμερα αυτό δείχνουν. Ακόμα όμως, κι αν μπορούμε να δημιουργήσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον κατάλληλο τρόπο, είναι γεγονό ότι δεν θα συμμετέχουν όλε οι χώρε μέλη εκεί. Άρα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στη Eurojust και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πρώτα απ' όλα να ενισχύσουμε τη συνεργασία μέσα στην ίδια τη Eurojust για να καταπολεμεί τέτοια εγκλήματα. Μόνο έτσι θα έχουμε αποτελέσματα και συμφωνώ επίσης για το ότι οι κοινέ ερευνητικέ ομάδες αποτελούν μια ευκαιρία για ενίσχυση της δουλειάς που ήδη κάνουν σήμερα επί τόπου. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε νέα όργανα. Πρέπει να προχωρήσουμε βέβαια, να φτιάξουμε επιτέλους αυτή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εισαγγελία. με μια προπόθεση όμως. Διότι αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορούμε να την έχουμε μόνο εφόσον υπάρχουν ενιαίες προδιαγραφές επί της διαδικασίας και επί του ποινικού δικαίου. Δουλεύουμε πάνω στο χάρτη πορείας, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Ελπίζω και εγώ το Συμβούλιο να έχει αποτελέσματα όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια προστασία υψηλού επίπεδου, όχι τελάχιστα μόνο που προβλέπονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά να μην μειωθούν οι προδιαγραφές σε σχέση με ό,τι ισχύει σε διάφορες χώρες μέλη. Και για την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Αγγελίας λοιπόν πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες διαδικαστικοί. Προς το παρόν δεν μου φαίνεται να είναι σαφές αυτό το Συμβούλιο να θέλει να βγάλει όλα τα διαδικαστικά, για μένα είναι κόκκινη γραμμή, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι σαφές ότι θα πρόκειται απλώς και μόνο για αναζήτηση ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να δεχτεί λοιπόν μια τέτοια πρόταση. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές από εμά. Τέλος. Προκειμένου να αποφύγουμε αυτό το forum shopping, την αναζήτηση δηλαδή ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας, πρέπει να Μην έχουμε Ευρωπαίο εισαγγελέα χωρίς δυνατότητες ε, αποκατάστασης επανόρθωσης. Κάτι πολύ βασικό για τις χώρες μέλη όπου δρά ο Ευρωπαίος Αγγελέας. Πρέπει και αυτή η απόφαση να ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει όλες τις διατάξεις που θα συμπεριλάβουμε εμείς στη νομική πράξη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερη ανεξαρτησία. Όχι. Αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δρά ως εποπτική αρχή. Και αυτή την ανεξαρτησία πρέπει να την ενισχύσουμε. Η καλύτερη δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ακριβώς να είναι ανεξάρτητη από εθνικές αρχές ε, για να αποφεύγεται η διαφθορά. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως θα πρέπει να αποτελεί το χώρο ο οποίος θα ελέγχει όλες τις πράξεις. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε όλα τα νομικά συστήματα τα οποία εμπλέκονται σε μία έρευνα. Στην ε, δικιά μου χώρα και σε άλλες χώρες όπου λαμβάνει η χώρα η διαδικασία αυτή. Αυτά σε σχέση με τις διατάξεις. Η διαδικασία λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν επιμείνουμε στις χώρες μέλη να συμφωνήσουν και να συμμορφώνονται σε ελάχιστες ε, προδιαγραφές ε, διαδικαστικές, τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ευχαριστώ. Βλέπω όντω ότι είναι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου οι παρεμβάσει των σχεδόν εισηγητών, αλλά θέλουν και άλλοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Άξελ Φώστορ. Παρακαλώ, Άξελ. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντ. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω αυτό που είπε και η κυρία Κάουφμαν και οι προλελήσαντες και ο κύριος ε, Άλμπρεχτ. Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα εργάζεται αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο κάθε κράτος ε, μέλος, διότι ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας ο οποίος θα έχει απλά μια ενισχυμένη θέση, είναι από μόνο του κάτι το αντιφατικό. Πρέπει λοιπόν αρχικά να δούμε ποια θα είναι η έκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Εισαγγελία. Δεν πιστεύω πως είναι, αρκε... αρκετό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και όπως είπε και ο Γιάνν Φιλιπ Άλμπρεχτ, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο ερώτημα του ποιος είναι ο αρμόδιος εισαγγελέα για την κάθε υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός ανεξάρτητος και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι δεν υπάρχει κώδικας ποινική δικονομίας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό. Επίσης υπάρχει και το πρόβλημα του forum shopping, όπως είπε και ο Γιάννη, τη ε, άγρας δικαστηρίου δηλαδή. Και εδώ πρέπει πιστεύω να σταθούμε στις επιμέρους αυτές οι λεπτομέρειες παρά να προσπαθούμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο σύνολό της. Υπάρχουν αυτά λοιπόν τα προβλήματα. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της ε, διασυνοριακής συνεργασίας της αρμοδιότητας του, της ε, κάθε χώρας και τις διαφορές στο δικαστικό σύστημα από χώρα σε χώρα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει μια τελείως διαφορετική διαδικασία που ακολουθείται. Υπάρχει μια ξεκάθαρη δομή και πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε μια πλήρη εναρμόνιση των δικαρδιστικών συστημάτων. Γι' αυτό λοιπόν ίσως βιαζόμαστε στην δημιουργία μιας ε, Ευρωπαϊκής εισαγγελία που να είναι, που να λειτουργεί έτσι. Χρειαζόμαστε και τις άλλες υπηρεσίες, χρειαζόμαστε τον Όλαφ και χρειάζεται επίσης να δαπανίσουμε πολύ περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να επιλύσουμε τα επιμέρους προβλήματα παρά να στεκόμαστε, να στεκόμαστε στη γενικότερη εικόνα, διότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συσταθεί σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Άξελ. Η κυρία Μέιρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι κατά της δημιουργίας μιας τέτοιας ε, εισαγγελία. Νομίζω ότι πρέπει το θέμα να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να παραμείνει. Για μένα δεν χρειάζεται μια τέτοια εισαγγελία και ακόμα και το θέμα των απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται για χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να είναι οι εθνικές αρχές οι οποίες να έχουν αυτήν την αρμοδιότητα. Κατόπιν τούτων, έχω και κάποιες ερωτήσεις. Η δικιά μου χώρα, η Ολλανδία, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτή η, αυτός ο ενιαίος ο χώρος ο δικαιοσύνης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποσαφηνίσετε περισσότερο. Και όσον αφορά τις ε, εθνικές αρμοδιότητες αυτού του ενιαίου χώρου επίσης. Θέλω να ξέρω και περισσότερα για τη συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα επ' αυτού. Τι θεωρούν οι διάφορες πλευρές όσον αφορά αυτή την έννοια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία λοιπόν βλέπει την δημιουργία αυτή σαν ένα βήμα για παρετέρω ενοποίηση της ε, ποινική διαδικασίας. Και ποιες χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για αυτήν την ενισχυμένη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η κυρία Σουίνιπερκ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει μέχρι τώρα. Έχω μια δήλωση να κάνω για να σας πω ποια είναι η θέση μας για το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να πούμε είναι ότι η έλεγχη ενός τέτοιου υπερκράτους είναι κάτι που γίνεται όλο και πιο σαφές. Και αν δούμε την δυνατότητα που έχει η Σουηδία να συμμορφωθεί με τον νόμο, μπορούμε να πούμε ότι οι Σουηδικές αρχές μπορούν κάλλιστα αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Οι Σουηδικές αρχές είναι απόλυτα ικανές χωρίς ε, καν να χρειάζεται αυτή η διασυνοριακή αντιμετώπιση, μπορούν κάλλιστα να αντιμετωπίσουν τέτοια εγκλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει βέβαια να βάλει τους δικούς της ανακριτές από τις Βρυξέλλες. Πίτερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα κάνω μια σύντομη και πιο γενική παρατήρηση για το θέμα αυτό, γιατί όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, στόχος του Συμβουλίου είναι να αποδυναμώσει την πρόταση και να περιορίσει ουσιαστικά τις εξουσίες ε, του Ευρωπαίου Ισαγγελέα, κάνοντας την υπηρεσία αυτή κάτι σαν την Eurojust με τη δυνατότητα αυτή εξουσιοδότηση εθνικών ε, εισαγγελέων. Έτσι οι χώρες μέλη είναι αυτές οι οποίες θα τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να αντιδρά σε αυτό που θέλουν οι πολίτες. Δεν μπορεί να αφήνουμε τις κυβερνήσεις να τα βρίσκουν μεταξύ τους ε, πίσω από κλειστές πόρτες. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και με μια πραγματικά αποτελεσματική υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εισηγηλίας. Πρέπει Λοιπόν, να λάβουμε υπόψη μας και να τροποποιήσουμε και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για την Όλαφ και την Eurojust για να αποφύγουμε επικαλύψεις και υπερβολική γραφειοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας πρέπει να ζητήσει μία εσωτερική προσωρινή έκθεση και να μπορέσουμε έτσι να πιέσουμε πολιτικά τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Πίτερ. Η Κατερίνα έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Και μετά εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Προεδρία για την παρουσίασή της και τους κοιόδης εισηγητές οι οποίοι έδειξαν πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει με την πρόταση αυτή. Πιστεύω ότι είναι όντως πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα και αυτό καταφάνηκε σήμερα. Κυρίως πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία και συμφωνώ με αυτό να έχουμε περισσότερη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία, όλες τις διαπραγματεύσεις όχι απλώς να ενημερωνόμαστε, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να παρέμβει με δικές του προτάσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς επειδή είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, παραμένουν σε κρεμότητα πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά την ίδια τη δομή, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τις εγγύησεις για την ανεξαρτησία της λειτουργίας αυτής και όσον αφορά διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Αλλά εγώ νομίζω ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να θέτουν υπό αμφισβήτηση τον ίδιο τον οργανισμό αυτό, την ίδια την υπηρεσία αυτή. Όχι, όλοι θέλουμε να βρούμε την καλύτερη, την ορθότερη λύση όσον αφορά τις δυσκολίες που σήμερα αναφέρθηκαν. Κάποιες χώρες θέλουν να συμμετέχουν και Κάποιες άλλες χώρες, όπως το ακούσαμε ήδη, μπορούν πολύ αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν ε, την ε, καταπάτηση αυτή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν στο μέλλον να παραδειγματιστούμε από τις χώρες αυτές και να μας βοηθήσουν να βρούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος να είναι ανεξάρτητος και να μπορεί να φέρει σε πέρα το ρόλο του. Η ενισχυμένη συνεργασία είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση στη συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτών και αυτό που είπα και πριν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και να συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Κλείνω τον κατάλογο μιλητών. Επόμενος είναι ο κύριος Λόπες Άγγιλαρ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλόντο. Πιστεύω κι εγώ ότι είναι σημαντικό κάθε φορά που αρχίζουμε μία συζήτηση για την διαδικαστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή ενός άρθρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό το οποίο προβλέπει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξανανοίγει ολόκληρη συζήτηση. Όχι μόνο για το πολιτικό επίπεδο, αλλά και για τις τεχνικές λεπτομέρειες της προπτικής δημιουργίας τελικά της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Οι τεχνικές λεπτομέρειες σίγουρα είναι δύσκολες, αλλά Νομίζω ότι είναι σωστό να επενθυμίσουμε εδώ ότι πρόκειται για ένα πολιτικό σώμα. Φυσικά και χρειάζεται πολλή δουλειά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι μόνο, αλλά και από το Συμβούλιο. Κάθε χώρα μέλη πρέπει να φροντίσει να προσφέρει ό,τι μπορεί σε αυτή αυτή την ε, προσπάθεια που είναι μοναδική στη φύση της. Δηλαδή πρέπει το κάθε κράτος μέλος να φροντίσει να διασφαλίσει και τις ε, διαδικαστικές διατάξεις αλλά και την ουσία. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό σώμα το οποίο έχει ως στόχο να καταπολεμήσει τη διασυνοριακή εγκληματικότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. κάτι το οποίο ξεπερνάει τις ε, αρμοδιότητες της διαφόρων ε, υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον νόμο είτε τις εθνικές είτε τις ευρωπαϊκές. Είναι κάτι διαφορετικό. Άρα μην ξεχνάμε το πολιτικό σκέλος. Γιατί φυσικά και καταλαβαίνω και πάντα το καταλάβαινα ότι υπάρχουν διαφορές διαδικαστικού τύπου όσον αφορά τα δικαιώματα. Ε, υπάρχουν διαφορές λοιπόν μεταξύ των χωρών όσον αφορά την αντιμετώπιση των ε, υπόπτων και κατηγορουμένων. Όντως είναι διαφορετικές οι σχετικές υπηρεσίες στις χώρες μας. Αλλά χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια τέτοια ευρωπαϊκή εισαγγελία ακριβώ για να ξεπεράσει τι αδυναμίε των υπηρεσιών αυτών που φροντίζουν για την επιβολή του νόμου στις χώρες μέλη ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο και να μην ξαναρχίζουμε να συζητάμε γι' αυτό. Φυσικά και υπάρχουν οι τεχνικές λεπτομέρειες που είναι περίπλοκες, που είναι δύσκολες, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό έρχεται σε ένα επόμενο στάδιο και θα ασχοληθούν με αυτές όταν φτάσει η ώρα οι χώρες μέλη. Όταν μιλάμε για τη διαδικασία όμως, το μήνυμα που πρέπει να στέλνουμε ότι είναι, είναι ότι είναι για καλό σκοπό που το άρθρο αυτό 86 αναφέρει Ήδη στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της ελευθερίας και δικαιοσύνης που αναφέρει τη δυνατότητα αυτή. Γι' αυτό θεωρώ τον αυτό μου υποχρεωμένο να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να μείνει στην πολιτική αρχή. Ότι δηλαδή πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσει την πρόταση αυτή και μάλιστα όσο γίνεται πιο γρήγορα για να δούμε να γίνεται πραγματικότητα αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Βόη, τελευταίο ομιλητή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο βασικό ερώτημα το οποίο ανέφερε και η σχεδόν κυρία Κάουφμαν. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δηλαδή πρέπει να γίνονται σεβαστά. Αυτό πιστεύω πως είναι αποφασιστική σημασίας και αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και την Κομισιόν αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές δηλαδή γιατί η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει τους ε, λόγους διακρίσεων και την απαγόρευση των διακρίσεων. Η Γερμανία έχει σχετική νομοθεσία και έχει ακολουθήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε όλα εκτός από αυτό ακριβώς το θέμα, το θέμα των ε, διακρίσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η οποία δεν λαμβάνει χώρα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες χώρες. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει κάποιος κατάλογος στον οποίο καταγράφονται αυτές οι περιπτώσεις διακρίσεων. Ή τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται μόνο εν μέρη σεβαστά. και τι δυνατότητα υπάρχει για να επιβληθούν στις χώρες αυτές ε, να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Ε, τι γίνεται με τις εκδόσεις πολιτών σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε τώρα στην εισηγήτρια, κυρία Μακοβέη. Και θέλω πραγματικά να ακούσω και τις απόψεις σε Συμβουλίου Επιτροπής. Ελπίζω να άκουσαν όλες αυτές τις εξαιρετικές παρεμβάσεις και να απαντήσουν στα συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Άκουσα με προσοχή τα όσα είπε ο Φερνάντο. Αλλά και οι σκιώδεις όλα τα μέλη μας έχουν ε, παρακολουθήσει εδώ και καιρό τις εξελίξεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ε, εδώ η ουσία του ζητήματος είναι οι διαφορές μεταξύ συστημάτων ε, δικαιοσύνης. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν πολλά πράγματα και να τα κάνουμε όλα σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο για μας. Επομένω. και μετά όσο ακούσαμε και από τον Φερνάντο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το εγχείρημα για το Κοινοβούλιο. Ε, δεν είναι επιφανειακό το έργο αυτό, γιατί έχουμε να κάνουμε ανταγωνιστικά συστήματα ποινική δικαιοσύνη ή τουλάχιστον διαφορετικά. Θέλω όμως να ξανακούσουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να απαντήσουν ε, στα συγκεκριμένα ερωτήματα που ακούστηκαν. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Μακοβέη και μετά Συμβούλιο και Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Συγγελία προβλέπεται στην συνθήκη. Δεύτερον, δεν μπορούμε να περιμένουμε τους ε, διαδικαστικούς νόμους ποινικού δικαίου για να θεσπίσουμε την Ευρωπαϊκή Συγγελία. Υπάρχει ανισομετρία στα εθνικά συστήματα. Ε, το ευρωπαϊκό ε, δικονομικό δίκαιο είναι ένα μακρόπνο σχέδιο, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τότε. Πρέπει να εγκαθιδρύσουμε την Ευρωπαϊκή Συγγελία. Επίσης, να επιθυμίσω στους συναδέλφους ότι για το 2013 η απάτη βάση του ελεγκτικού συνεδρίου ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Δις, μάλλον. Ε, σε επίπεδο διαφθορά αφορά τα 20 δις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, πολλά χρήματα χάνονται, πολλοί εγκληματίες ξεφεύγουν από τα χέρια του νόμου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό και έχει εγγραφεί στη συνθήκη όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία έρευνα στην Ιταλία, ακολουθούμε το Ιταλικό σύστημα. Στη Γερμανία μετά έχουμε την Ευρωπαϊκή Συγγελία, ακολουθείται μετά το Γερμανικό Δίκαιο. Και στο τέλος της έρευνας, όταν ο ευρωπαϊκός Αγγελίας θα αποφασίσει πού θα εκδικαστεί η απόφαση, και εκεί θα υπάρξει η δίωξη, τότε σε αυτό το δικαστήριο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ε, συλλεγεί κατά τη διάρκεια της ε, έρευνας θα αναγνωριστούν. Γι' αυτό γίνεται η έρευνα μέχρι το τέλος και μετά αναλαμβάνουν τα δικαστήρια. Τώρα τι έχουμε. Ο ΛΑΦ κάνει τη διοικητική έρευνα, στέλνει ε, στα, στις αθηνικές αρχές ό,τι έχει και πάνω από το ίμιση των ερευνών δεν συνεχίζονται στα κράτη-μέλη. Έπειτα. Σε κάποια τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Αλλού όμως, σε αλλα κρατημέλη δεν ανακτώνται τα χρήματα των φορολογουμένων και θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι όλοι αυτοί οι πόροι πρέπει να ανακτώνται. Υπάρχουν και αυτά τα κράτη μέλη που τα πάνε πάρα πολύ καλά λοιπόν, αλλά δεν μπορούν να λάβουν και όλο το βάρος για όλα τα κράτη-μέλη. Αν υπάρχει λοιπόν βούληση μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί όλα αυτό το παρόν κάνει τα διοικητικά. Ε, η δικαστική συνεργασία Europol Eurojust είναι κάτι το διαφορετικό. Η Ευρωπαϊκή Συγγελία θα αναλάβει λοιπόν ένα ξεχωριστό μοναδικό καθήκον, να ξεκινά δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος μια έρευνα κατά τυχαίο τρόπο να γίνεται ο καταμερισμός των ερευνών, να υπάρχουν έρευνες σε άλλα κράτη-μέλη για να υπάρχει αμεροληψία και όλα τα αποτελεστικά στοιχεία να αναγνωρίζονται από το δικαστήριο που ε, θα εκδικάζει την ε, υπόθεση. Αυτά θέλουμε να κάνουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τα όσα είπε η κυρία Μακοβέη. Έχουμε και εμείς τον ίδιο σκοπό. Θέλουμε ένα, μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και πολύ ανεξάρτητη εισαγγελία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε κατόπιν και του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου να ε, γίνει ακόμα πιο ανεξάρτητος αυτός ε, ο οργανισμός με την εκλογή του Ευρωπαίου Εισαγγελέα το τώρα δυνατόν. Στη συνέχεια θέλω να απαντήσω και στον κύριο Μισελ που ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο θέλουν να προχωρήσουν το στενότερο δυνατόν για να υπάρξει ταχεία υιοθέτηση του σχεδίου κανονισμού. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι υπάρχει κάτι τέτοιο για την Επιτροπή. Από πλευρά Συμβουλίου μπορώ να μιλήσω για την δική μας βούληση, της Προεδρίας δηλαδή, ε, και δεν μπορώ να προδικάσω τη θέση των υπολείπων κρατών μελών. Τώρα, να σχολιάσω τα όσα είπαν η κυρία Κάουφμαν και ο κύριο Άλμπρεχτ. Δεν ήμουν αρκετά σαφή, μάλλον προηγουμένω. Είπα ότι θέλουμε να διαγράψουμε ε, διατάξει επί τη διαδικασία, αλλά μάλλον δεν τα είπα εγώ ξεκάθαρα. Θέλουμε ένα εύρωστο, ισχυρό σύστημα προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Δεν θέλουν καθόλου τη διαγραφή του. Το υφιστάμενο σύστημα, και μάλιστα σε αυτό αφιερωθήκαμε και με αυτό ασχοληθήκαμε στο Συμβούλιο στο Μιλάνο, έπρεπε να δείτε το επίπεδο φιλοδοξίας για την ε, προστασία ε, των οικονομικών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο που σημαίνει ότι οτιδήποτε έχει υιοθετηθεί, έχει υιοθετηθεί και επιπλέον θα έρθουν τα εθνικά μέτρα η Ιταλική Προεδρία έχει λάβει δύο προτάσεις που είχαν τεθεί επιτάπητος από τον περασμένο Δεκέμβριο στο Συμβούλιο και τα έχουμε προωθήσει. Λογικά τον Δεκέμβριο θα οριστικοποιηθεί η οδηγία ε, για την ε, τεκμήριο της αθωότητας. Θέλουμε να ε, ενταχθεί Θεωρούμε ότι πρόκειται για θεμελιώδε δικαίωμα. Θέλουμε λοιπόν να ενταχθεί και στην πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χαιρετίζω και την ε, πρόσκληση τη ε, κυρία ε, Κάουφμαν. Σίγουρα και το Δεκέμβριο θα δημοσιευθούν αυτά, γιατί θα έχουμε, πλέον, θα έχουμε περάσει στους υπουργούς και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Τώρα έχουμε τον βασικό πυρήνα της πρότασης και ελπίζουμε να διαβιβαστεί και στο ε, Κοινοβούλιο. θέσατε ένα ερώτημα για το αν θα έχουμε σε εισαγγελία. Είναι το αρχικό σύστημα. Δεν λέμε ότι γενικά κάθε τρία χρόνια θα υπάρχει αναλλαγή. Στην αρχή, όπως ισχύει και με άλλους δικαστικούς οργανισμούς και φορείς, όταν υπάρχει ένας, ε, συστήνεται ένας φορέας μετά περνάνε κάποια χρόνια και μετά φεύγουν όλοι την ίδια στιγμή. Γι' αυτό έχουμε ένα σύστημα τέτοια αναλλαγή ε, κάθε τρία χρόνια. Αλλά μετά κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτή, αυτό το σύστημα. Δεν πρέπει να μας απασχολεί και να μας προβληματίζει λοιπόν. Για τα ερώτημα της Bundestag, ε, για τους επικεφαλής εισαγγελείς, πρέπει να το προτείνουμε αυτό στους ε, υπουργούς, ένα πιο αποτελεσματικό δίκτυο εξασφάλισης της ανεξαρτησίας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε αυτό το στάδιο εξετάζουμε ε, την ιδέα μιας ε, κριτικής επιτροπής βάσει του συστήματος που ακολουθείται και στο δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και την εκλογή των δικαστών με μια ανοιχτή διαδικασία ανοιχτή προ όλου, ε, Θα προτείνετε λοιπόν, θα επιλέγετε μάλλον ένας ε, σύντομος κατάλογος που θα υποβάλλεται προ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που θα συναποφασίζουν. Όπω ε, ισχύει και με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Προστασία Δεδομένων. Για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων με τη Eurojust και άλλους φορείς, ειλικρινά δεν μπορώ να σας απαντήσω πλήρως αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε ακόμα εξετάσει αυτές τις διατάξεις. Πιστεύω όμω ότι χρειαζόμαστε ένα εξαιρετικά σαφέ κείμενο για την πρόταση οδηγίας, για την προστασία οικονομικών συμφερόντων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας συνδέεται στενά με ε, τον ορισμό αυτών που προβλέπεται στην οδηγία ε, που προανέφερα και η κυρία Γκρέσλε και ο κύριος Λόπες Κίγια έχουν ε, οριστεί στην ομάδα που ξεκινά τον ε, άτυπο τριμερή διάλογο και συνεχίζουμε ταχύτατα για την υιοθέτηση μιας οδηγίας που θα περιλαμβάνει και σαφείς ορισμούς. Αν έχουμε σαφείς ορισμούς στην οδηγία, θα έχουμε και σαφή εντολή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ποια ακριβώς αδικήματα υπόκειται στο πεδίο αρμοδιοτήτων και ποια όχι. Μετά, νομίζω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα είναι κρίσιμη σημασία θέμα. Ο διάλογος ε, και οι επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελία και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών όπως η Eurojust απαιτούν ένα σύστημα με αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και ιδίω ό,τι αφορά τη Eurojust, ε, θεωρούμε ότι ο ρόλος της είναι ουσιαστική σημασία για να διασφαλίσει συνεργασία μεταξύ ε, ΕΠΟ και τρίτων χωρών. Όχι μόνο τρίτων χωρών, γιατί ακούσαμε ότι δεν θα συμμετέχουν και όλα τα κρατημέλη. Ένα μάλιστα εξαιρείται βάσει του ε, κεφαλαίου 5 της συνθήκης. Θα δούμε για τα υπόλοιπα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η Eurojust σίγουρα θα διαδραματίσει πολύ ουσιαστικό ρόλο. Για το κόστος, να το αφήσουμε τα χαρά στο συνάδελφο τη Επιτροπής να το απαντήσει αυτό. Ήδη έχει τεθεί αυτό το ζήτημα όμω. Ποιο ακριβώ θα αναλάβει το κόστο τη Ευρωπαϊκή Αγγελία όταν περάσουμε σε αυτό το σύστημα του συλλογικού οργάνου. Τα κράτη-μέλη θα το αναλάβουν ή το κόστος θα καλυφθεί από τον κοινοτικό προπολογισμό. Είναι όμως κάτι το οποίο έχει τεθεί επιτάπητος. Να περάσω τώρα στα όσα είπε η κυρία Μέιερ. Ενιαίος νομικός χώρος. Είναι μια ωραία έκφραση, αλλά είναι και μια ιδέα. Προσπάθησα να την ε, παρουσιάσω προηγουμένως. Ε, ένας χώρος όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να συλλέξει στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία, ε, να εφαρμόζει ερευνητικά μέτρα χωρίς να έχει αντιμέτωπη με σύνορα ουσιαστικά. Να μην ξεχνάμε λοιπόν όμως ότι υπάρχει ένα ε, σύστημα εξουσιοδοτήσεων, δηλαδή θα υπάρχει δράση σε εθνικό επίπεδο με τις τοπικές ε, αρχές επιβολής του νόμου. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα υπάρχει απόλυτο σεβασμός προς το εθνικό σύστημα, γιατί θα έχουμε ένα αποκεντρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα αν θα έχουμε έναν ε, ευρωπαϊκό κώδικα ποινικού δικαίου, όχι. Απλώς σε αυτό το στάδιο προσπαθούμε να εναρμονίσουμε ε, τον εσωτερικό κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά η δίκη πάντα θα γίνεται ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου, όπως γίνεται και σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα παρουσιάζει όλα τα στοιχεία στο Εθνικό Δικαστήριο και εκεί θα συνεχίζεται η διαδικασία. Και τέλος, να απαντήσω και στον κύριο Βόιτ για τις εκδόσεις. Ήδη υπό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ευρωπαϊκού Εντάλματος προβλέπεται η έκδοση υπηκών ενός κράτους μέλους προς άλλο. Και εδώ το σύστημα δεν είναι πολύ διαφορετικό, ακόμα το συζητάμε αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ζητήσει από δικαστική αρχή να εκδώσει ε, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Ουσιαστικά μιλάμε για αυτά που ήδη ισχύουν από το 2002. Ελπίζω να απάντησα στα περισσότερα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε όσα είπε ο συνάδελφος από το Συμβούλιο, αλλά να πω καταρχάς ότι μας χαροποιεί που ακούμε τόσο θετικά λόγια για τη δημιουργία αυτού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής εισαγγελία και για το ότι συμφωνείτε με τις ε, κόκκινες γραμμές που έχουμε θέσει και εμείς από ό,τι φάνηκε από τα σχόλια των ε, εισηγητών, των σκηνοδών εισηγητών και των υπόλοιπων ευρωβουλευτών της Επιτροπής αυτής. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι με χαρά μας θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας για την συνέχιση αυτού του τόσο σημαντικού θέματος. Αναφέρθηκαν πάρα πολλά σημαντικά θέματα. Ένα από αυτά είναι η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Eurojust και την Olaf. Και φυσικά πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα του κόστου, το οποίο ήδη αναφέρθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκεφτεί πολύ για το πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα και μπορώ να σας πω ότι σε περίπτωση αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής εισαγγελία, τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν πλέον την ε, εθνική αρμοδιότητα για κάποια υπόθεση και η Eurojust δεν θα μπορεί να συντονίσει την ε, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Από την άλλη βέβαια, σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό. Φυσικά και θα μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε. Και εδώ να επιβεβαιώσω και εγώ αυτό που είπε το Συμβούλιο για την συνεργασία με τρίτα κράτη, το οποίο προβλέπεται στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελία. Τώρα για το ζήτημα του κόστους. Να σας πω ότι φυσικά και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος. Αν δείτε τους υπολογισμούς μας θα ε, δείτε ότι κάποιες εργασίες θα αφαιρεθούν από την Όλαφ και από την Eurojust για να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι λοιπόν δεν θα αυξηθεί πολύ το κόστος. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι υπολογισμοί που δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη. Ο μισθός, για παράδειγμα, των Ευρωπαίων εισαγγελέων θα γίνεται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα και θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Τώρα, όσον αφορά τις ε, εγγύησεις για τα νομικά δικαιώματα, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύουμε, να υπάρχουν αυτά τα δικονομικά δικαιώματα στο κεκτημένο. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί σωστά μόνο εφόσον γίνονται σεβαστά αυτά τα δικονομικά δικαιώματα σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Και θα το αφήσω εδώ το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Θα προχωρήσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης και θα ήθελα όμως εδώ να ζητήσω στον Γιάννη Μπρέχτη να πάρει τη θέση του Προέδρου και να συνεχίσει εκείνος τη συνεδρίαση. <laughs> brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. Okay, we can just start. Mm-hmm. Okay, dear colleague. Αγαπητοί συνάδελφοι, για το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης έχουμε αφήσει την ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης. Έχουμε συντάξει μια γνωμοδότηση για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Η συγκήτρια είναι η κυρία Μόνικα Μάκοβέη επίσης. Και επίσης θα έχουμε, και την, συνέχ... θα έχουμε την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης. Θα δώσω το λόγο αμέσως στη Μόνικα Μακοβέη για να μας κάνει την εισαγωγή στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Το 2013 καταγράφηκαν πάνω από 15.000 παρατυπίες. Και από αυτές τις 15.000 περίπου 1.600 περιπτώσεις αφορούσαν περιπτώσεις απάτης που κόστησαν περίπου 309 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι η συγγήτρια του ΕΛΚΑ από το 2009 για αυτό το θέμα και παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις διότι πρόκειται για χρήματα των φορολογούμενων. Έχουν γίνει πάρα πολλές αναλύσεις στα, στις παρατυπίες αυτές. Παρακολουθούμε λοιπόν τις, την υπηρεσία συντονισμού καταπολέμησης της απάτης που γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος Ηρακλής. Εκτός από συγγήτρια της Επιτροπής Ελίμπε στο θέμα αυτό, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ο κανονισμός αυτός για το ΕΛΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικά μέσα καταπολέμησης της απάτης στο ποινικό δίκαιο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δοθούν σαφείς ορισμοί για τα ποινικά αδικήματα, να δοθούν σαφείς ορισμοί για τις ελάχιστες και μέγιστες ε, ποινές και σαφείς κανόνες για τους ε, περιορισμούς που υπάρχουν. Επίσης, πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη υπηρεσία που θα οδηγεί στη δικαιοσύνη τους ε, παραβάτες, σεβόμενη τα, τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διαδικασία των εισαγγελέων θα πρέπει να είναι διάφανοι και οι εισαγγελίε θα πρέπει να επιλέγονται μετά από διαβουλεύσει με τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτό συνδέεται και με την πρόληψη και ανάκτηση των χαμένων πόρων της Ένωσης. Επίσης, η θέση του Κοινοβουλίου πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα πλαίσια της συνεργασίας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συνένεσης και σε εθνικό επίπεδο και μετά σε θεσμικό επίπεδο. Τώρα, θέλω να τονίσω την ε, σημασία ορισμένων μέσων όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Περικλής 2020 και το πρόγραμμα Ηρακλής 3 για τους, ε, την ανάκτηση οικονομικών πόρων. Αυτά συνοπτικά από εμένα. Ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και με χαρά μου να συμπεριλάβω τα σχόλιά τους στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές και πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι συγητής της ΛΥΜΠΕ για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. σε σχέση με το ποινικό δίκαιο. Γι' αυτό θα ήθελα να δούμε το περιεχόμενο και το νόημα της γνωμοδότησης αυτής και να πω ότι συμφωνώ με όλα τα επιμέρους στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στη γνωμοδότηση αυτή. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή που δείχνει τη σημασία που έχει η ολοκλήρωση της οδηγίας προκειμένου να μπορέσουμε καλύτερα να καταπολεμήσουμε την απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε για τους τρεμερείς διαλόγους που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σας ε, υπενθυμίζω πως ναι, χρειάζεται σαφήνεια όσον αφορά τον ορισμό των αδικημάτων και των εγκλημάτων που αποτελούν απειλή στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ε, που πρόκειται για κατάχρηση, διαφθορά, άμεση-έμεση και συμπεριφορά των αξιωματούχων, που και αυτό εξακολουθεί να είναι ένα θέμα σε κρεμότητα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα καταλήξουμε σε ξεκάθαρους ορισμούς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τους συμβιβασμούς επίσης. Υπάρχει το θέμα της παραγραφής, υπάρχουν διαφορές στις προθεσμίες ανάμεσα στις χώρες μέλη. Υπάρχουν διαφορές στην εθνική νομοθεσία. Αυτό συμβαίνει σε πολλά θέματα. Για το κατά πόσο θα συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ή όχι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να παραμείνει αυτό το θέμα. Αυτή ήταν η θέση μας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε εδώ. Όσον αφορά τον τριμερή διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα, επίσης αυτό υποστηρίξαμε. Τώρα έρχομαι στα άλλα θεσμικά όργανα. Eurojust, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Όλαφ. Γιατί και Όλαφ αυτή τη δουλειά κάνει. Προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται και συνδέονται τα όργανα αυτά μεταξύ τους. Να μην καταλήξουμε σε ένα λαβύρινθο και χαθούμε εκεί, ούτε να δίνουμε την εντύπωση ότι προσθέτουμε οργανισμούς όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα το θέμα να γίνει πιο περίπλοκο και να μην καταφέρουμε τελικά να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της απάτης. Αυτά τα θέματα βέβαια έχουν να κάνουν με το ίδιο το ποινικό δίκαιο. Γιατί το ποινικό δίκαιο διαφέρει. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει και τη διαφορά στο θέμα. Γι' αυτό και συμφωνώ με τόσα αναφέρει η γνωμοδότηση που άκουσα από την εισηγήτρια την κυρία Μακοβέη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ενημέρωση που μας έδωσε. Όντως θα ήταν καλό να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό όμως που διαπιστώνω είναι ότι μελετώντας το έγγραφο υπάρχει σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Και συμμερίζομαι επίσης την ιδέα που λέω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή ε, τα μέσα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες μέλη και την Ένωση. Συμφωνώ συνεπώς απόλυτα με τη δημιουργία αυτού, του, αυτής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα προσθεθεί στα όργανα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να διευκρινιστούν διάφορα πράγματα όσον αφορά την παραγραφή. Το ανέφερε και ο κύριος Λόπες Άκυλαρ εξάλλου. Ή όλο το θέμα των μηχανισμών που έχουν να κάνουν με την κοινοποίηση και την διαχείριση των υπονιών για απάτη. Και εδώ λοιπόν πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά περισσότερο σε βάθος. Πάντα με στόχο να δημιουργήσουμε τα όργανα εκείνα τα οποία θα είναι πραγματικά αποτελεσματικά και θα μας επιτρέπουν να ελέγξουμε καλύτερα την κατάσταση και να καταπολεμήσουμε καλύτερα και να προλάβουμε μάλιστα τις απάτες όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. σε ευχαριστούμε. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, τότε παρακαλώ να πω ότι συμφωνώ και εγώ με το ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και θα δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Μακοβέη για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Συμφωνούμε. Απλώς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η γραμματεία θα σας ενημερώσει όταν θα είναι έτοιμες οι μεταφράσεις όλες τις γλώσσες. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 8 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία της νομοδότησης θα λάβει χώρα στην Επιτροπή μας λίγο 8 Ιανουαρίου. Έτσι η Επιτροπή, Προπολογισ... η Επιτροπή Προπολογισμών μπορεί να τα ελέξει. Έληξη συνεδρίαση. Α, συγγνώμη. Να σας πω και για την επόμενη συνεδρίαση, λέει ο Πρόεδρος. 2 Δεκεμβρίου, 11 με 12 και 30. Θα είναι μια κοινή συνεδρίαση, συνεδρίαση, FAM-LIBE, με την συντονίστρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση εμπορία ανθρώπων, την Μύρια Βασιλιάδου, όσον αφορά τη στρατηγική 2012-2016, στην αίθουσα Γιάν 6Q2. Και μετά έχουμε προβλέψει συνεδρίαση στις 3 Δεκεμβρίου, 9 με 12 και 30 και 3 με 6,5 και 4 Δεκεμβρίου, 9 με 12,5 και 3 με 6,5. Σας ευχαριστώ και καλό απόγευμα. Whatever.